Βάσει του άρθρου 216 εδάφιο 4 σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει καμία αίτηση για να εφαρμοστεί στις ψηφοφορίες στο διορθωτικό που ανακοινώθηκε χθε στις 12. Οπότε θεωρούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση για το διευθυντικό εγκρίνεται. Περνάμε στις ψηφοφορίες.